πάντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ερυθρέα συγκεκριμένα οι περιπτώσει των Αμπούνε Αντώνιου και Ντάβιτ Ισακ. Οι συντάκτε πρώτη, η κυρία Βαλέρο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να σας πω και τον Ντέβιτ Ίσακ που είναι Σουηδός υπήκος και φυλακίστηκε χωρίς δίκη στην ε, Ερυθρέα στη συνέχεια των επιθέσεων του δικαστήριου στην ε, Αμερική φημώθηκε ο τύπος και 11 και περισσότεροι δημοσιογράφοι χωρίς δίκη φυλακίστηκαν. Συνεχίζεται μόνο η καταστολή παρά την διεθνή πίεση. Στη Σουηδία υπάρχει κίνημα για την απελευθερωσή του και το 2010 είχαμε μια έκθεση σύμφωνα με την οποία ή τέλο πάντων κάποια αναφορά που έλεγε ότι κρατείται σε υπόγειο υπό συνθήκες άθλιες ούτε νερό δεν έχει αλλά πάντως το πιο σημαντικό είναι ότι με αξιόπιστε πηγές βεβαιώνεται ότι ζει φυλακίστηκε με άλλους που δεν έχουν δικαίωμα σε δίκη. Υποφέρει αυτός και η οικογένειά του και γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι σημαντικό τον λόγο ψήφισμα. Ευχαριστούμε. Πώς; 1,5 λεπτό. Thank you, Madam Chair. Ε, we as a group... Ναι, κύριε Πρόεδρε, εμείς ως σοσιαλδημοκράτε είμαστε προσιλωμένοι στο έργο μας ούτω ώστε να γίνονται σεβαστά όλα τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και για αυτό το λόγο και προωθήσαμε αυτό το ψήφισμα. Βλέπουμε να κλιμακώνεται η βία κατά ακτιβιστών και δημοσιογράφων σε όλο τον κόσμο. Έχουν περάσει από τότε 16 χρόνια. Ο Ίσακ και άλλοι δημοκράτες και ε, ακτιβιστές είναι φυλακισμένοι είναι σύμβολο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ευφυΐας του τύπου. Αλλά για πολλού είναι πάνω από ένα σύμβολο πίσω στην πατρίδα, στην Σουηδία, όπου λείπει από την οικογένειά του. Τους λείπει πολύ και αυτός και οι άλλοι. Και μετά από αυτά τα 16 χρόνια ας μπορούσαμε τουλάχιστον να ακούσουμε ένα μήνυμα από το στόμα του. Ακούστε μας λέμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί το Κοινοβούλιο Πανελλημένα έχει πει ότι δεν είναι δυνατόν να κάνουμε αναπτυξιακή βοήθεια με χώρες που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και που δεν προτίθενται να απελευθερώσουν τον Ίζερ. Ήδη υπάρχει μια συμφωνία 200 εκατομμύριων ευρώ. Όμως με ένα απλό κείμενο, αν δώσουμε τα χρήματα, τα πράγματα θα είναι μία από τα ίδια. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε τόσο ώστε να υπάρξει δημοκρατία. Να μην στείλουμε ούτε μια δεκάρα σε αυτό το καθεστώς. Να μην ξεχνούμε, θα πρέπει να κλείσετε λέει πρόεδρος. Δεν θέλουμε να τους προδώσουμε και να τους εγκαταλείψουμε λέει η ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ. Και η επόμενη συγγετρία, η κυρία Βίξτρομ, επίσης για μισή λεπτό έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Πρόκειται για έναν ε, δημοσιογράφο από της και της Σουηδίας, ο οποίος ε, φυλακίστηκε για 15 χρόνια χωρίς να έχει οποιαδήποτε επαφή με την οικογένειά του, χωρίς να έχει περάσει από δικαστική αγωγή. Ντάβιτ Ιζακ, το όνομά του, έχει επιδείξει τρομερό θάρρος ως δημοσιογράφος έχει πραγματικά θέσει την ίδια τη ζωή του σε κίνδυνο για να μιλήσει για, τα, για τις ιστορίες ε, των ανθρώπων. Ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τώρα είναι στη φυλακή. Και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας τα οποία διαπράττει η Ερυθρέα δεν μπορούν να συνεχιστούν. Πρέπει επιτέλους η Σουηδική Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσουν τα μέσα που έχουν στην ε, διάθεσή τους για να ασκήσουν πίεση στην Ερυθρέα. Θα πρέπει να απαγορευτεί απαγορευτούν τα ταξίδια σε ό,τι αφορά την Ερυθρέα να φροντίσουμε για τους πολίτες με ευρωπαϊκή ηθαγένεια που βρίσκονται στην Ερυθρέα και θα πρέπει επιτέλους να εξασφαλίσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα τηρούνται στην Ερυθρέα να προασπίσουμε την ε, δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή είναι η πιο σημαντική μας δουλειά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην επικρατειά μας και σε όλο τον κόσμο. Και θα πρέπει λοιπόν να καταγγείλουμε όλα αυτά τα εγκλήματα και ο Ντάβιντ Ιζάκ έχει αγωνιστεί υπέρ τη Δημοκρατία και πιστεύω ότι αξίζει να είναι υποψηφίο για το βραβείο Ζαχάροφ. Είναι λοιπόν δική μα ευθύνη πλέον να υψώσουμε τη δική μα φωνή για να α, μιλήσουμε για τον Ντάβιντ Ιζάκ. Κυρία Βέξτρομ, έχετε μια μπλε κάρτα από την ε, κυρία Γκόμε. Την δέχεστε, κυρία Γκόμε, έχετε 30 δεύτερα στη διάθεσή σα. Συνάδελφε Βίξτρομ, είπατε ότι ο Ντάβιτ Ιζάκ ήταν ο μοναδικός ε, φυλακισμένος συνείδηση στην Ευρώπη. Έχετε υπόψη σας ότι αυτό δεν αληθεύει και ότι υπάρχει ο Βρετανός Αιθιόπιος πολίτης Τσίκε, ο οποίος επίσης ε, έχει απαχθεί και φυλακιστεί. όσο και να θέλω να επιδείξω αλληλεγγύη προ εσά για την ε, μοίρα του Νταβίτ Ιζάκ δεν στέκει το να λέμε ότι είναι ο μόνο. Η κυρία Βίξτρομ έχει 30 δεύτερα για την απάντηση Αγαπητοί συνέδελφε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο να τσακωνόμαστε γι' αυτό. Ο Νταβίτ Ιζάκ για πάρα πολύ καιρό 15-16 χρόνια τώρα κοντά. Είναι φυλακισμένος λόγω αντιρρησίας συνείδησης. Ε, αν υπάρχουν και άλλοι, προφανώς ε, το δέχομαι. Ε, ας αγωνιστούμε για όλους τους. Και αν υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι φυλακισμένοι, σημαίνει ότι δεν έχουμε εργοποιηθεί επαρκώς. Ευχαριστώ ο κύριος Τάνοκ τώρα για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το Καθεστώ ε, τη ε, Ερυθρέα οδηγεί στην καταστροφή τη ευημερία της χώρας αυτή από τότε που απέκτησε το 1991 την εξαρτησία της από την Αιθιοπία. Πρέπει να δούμε ολόκληρη τη διπλωματική εικόνα. Επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε δύο κρατούμενους, τον Δαβερή Σάκα και τον Πατριάρχη Αντώνιο, ο οποίος ε, είναι Πατριάρχη τη Ορθόδοξη Εκκλησία εκεί. Και αυτοί είναι στη φυλακή και δημοσιογράφοι εδώ και 10 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, ο Ντάβιτ Ισακ είναι κάποιος για τον οποίο δεν έχουμε νέα από το 2005. Όλα αυτά δείχνουν Πώ προχωράει το ολοκληρωτικό καθεστώ τη Ερυθρέα που οδηγεί σε χιλιάδε ανθρώπου να φεύγουν για να αποφύγουν τι καθημερινέ Εξήντα 60.000 είναι ανά το κόσμο. Είναι η ένατη μεγαλύτερη χώρα προσφύγων ανά το κόσμο όταν μιλάμε για μια χώρα για 6 εκατομμύρια, έτσι. Οπότε ζητάω από το Σώμα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσω διαβουλεύσει βάσει του άρθρου 96 τη συνθήκη του Κοτονού. Είναι κάτι που το λέω εδώ και έξι χρόνια και το ξαναλέω και τώρα. Ευχαριστούμε. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Μαρή Κριστίνε Βερζιά. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ο Ταβίτη Ζάκ αποτελεί ένα σύμβολο. Το Σεπτέμβριο του 2001 μαζί με άλλους δεκάδες συνελήφθη και μπήκε στη φυλακή επειδή αντιδρούσα στη δικτατορία. Δεν υπάρχει ελεύθερος τύπος εδώ και 7 χρόνια. Ο Αμπουλή Αντώνιος, ο Πατριάρχης Ορθόδοξης Εκκλησίας, είναι άλλο ένα σύμβολο. Το 2016 κρατήθηκε γιατί δεν δέχτηκε να αφορήσει αυτούς οι οποίοι δεν θέλανε Διακόπτη η Πρόεδρος. Μια στιγμή. Ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν έχω ε, μετάφραση στα τσέχικα, λέει ο μιλητής. Δεν ξέρω αν λειτουργεί. Τώρα λειτουργεί από ό,τι φαίνεται. Κυρία Βερζιά, αρχίζει ο χρόνος σας ε, με 20-25 λεπτά που σας δίνουμε έτσι, 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ, γιατί όντως... Ναι. Λοιπόν, πρέπει να ξαναβρω το νήμα. Πού ήμουνα, τι έλεγα. Λοιπόν, ξαναρχίζω την πρόταση, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, και να δείξετε κάποια κατανόηση, παρακαλώ. Έλεγα λοιπόν ότι του τελευταίου μήνε χειροτερεύουν τα πράγματα. Ο δικό εισηγητή του ΟΗΕ μιλάει για συστηματικέ παραβιάσει και γενικευμένε που μπορεί να αποτελούν εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα. Και αυτή ακριβώ τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει να κάνει εταίρο τη την Ερυθρέα σε ένα πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Ένωση με 46 εκατομμύρια συν 5 εκατομμύρια μέσω του προγράμματο ΡΟΚ, το οποίο έχει να κάνει με την κατάρτιση των ε, συνοριοφυλάκων και της αστυνομίας. Δεν πρόκειται όμως ο λαός της Ερυθρέας να υποφεληθεί από τα κονδύλια αυτά. Είναι αδύνατο σε αυτή τη χώρα να κάνει κανείς οτιδήποτε χωρίς να περάσει προηγουμένως από την κυβέρνηση. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Θα φύγουν κι άλλοι ε, πολίτες της Ερυθρέας προς άλλες χώρες. Τι θα γίνει με αυτό το καθεστώ στο οποίο οφείλεται τελικά η μετανάστευση. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Τελευταίο από του συζητητέ, ο κύριο Λαχθέσον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ερυθρέα είναι μία από τις πιο άτακτες δικτατορίες στον κόσμο. Ο πρόεδρος της ΑΕΦ ε, έχει εφαρμόσει το καθεστώς του φόβου με τις εξαιρετικές καταχρήσεις κατά των ιδιών πολιτών του και οι εγκληματικές πράξεις είναι πραγματικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Έχει φυλακίσει τουλάχιστον 10.000 πολιτικούς αντιφρανούντες. Σήμερα λοιπόν τονίζουμε δύο από τους ε, αντιφρένοντες αυτούς δύο αθώα άτομα τα οποία έχουν δει τη ζωή τους να καταστρέφεται. Ας μην σταματήσουμε ποτέ τον αγώνα για τον ε, Ίζα και τον Αντώνιο, να μην ξεχνάμε ποτέ το απαράμιλο θάρρος τους. Τρία μέτρα λοιπόν είναι σήμερα απαραίτητα. Καταρχάς ε, η Ερυθρέα θα πρέπει να λαμβάνει αρρωγή με αυστηρή αιρεσιμότητα Οφιόρκη και οι πατριώνε ότι θα πρέπει να διωχθούν για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Και ο μεγάλος λαός της Ερυθρέας αξίζει να ζει με ελευθερία. Έχουμε ευθύνη να τους βοηθήσουμε για να είναι πιο λαμπρό το μέλλον τους. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Και τώρα να περάσουμε σε δύο ομιλητές από πολιτικές ομάδες. Ο κ. Τσεκόφσκι έχει 30 δεύτερα στη διάθεσή του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να πω ότι η κατάσταση στην Ερυθρέα είναι δραματική εδώ και πολύ καιρό. Και αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερω είναι το πολιτικό περιβάλλον. Γιατί η χώρα δεν ε, τηρεί τι διεθνεί συμφωνίε. Δεν υπάρχει κράτο δικαίου, δεν υπάρχει ανεξάρτητο δικαστικό σώμα, δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει κράτο δικαίου. Και για μένα όλα αυτά καταδεικνύουν ότι πρόκειται για το χειρότερο αυταρχικό καθεστώ στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν προσυπογράφω απόλυτα στην προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι πεπισμένο ότι θα πρέπει ακόμα και πιο αυστηρέ κυρώσει να επιβάλλουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και πραγματικά τα καταφέρατε σε 30 δεύτερα να μιλήσετε. Ευχαριστώ από το ΕΛΚ ήταν ο κ. Τσεκόσκιτ και τώρα από Σοσιαλιστές και Δημοκράτες η κυρία Γκούτελαντ. Fru talman, den här klockan visar den stulna tiden ifrån David Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εδώ και 16 χρόνια είναι φυλακισμένο ο Ντέβιτ Ιζακ. 16 χρόνια βεβαιότητα για του αγαπημένου του, για την οικογένειά του. Ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στην κυβέρνηση της Ερυθρέας. Η Ερυθρέα θα πρέπει να απελευθερώσει άμεσα τον Δαβίδ Ιζάκ, να λάβει νομική αραγή και δεν θέλουμε άλλα λόγια, θέλουμε πράξεις. Θα πρέπει να μάθουμε κατά πόσο είναι σε καλή υγεία και οι πολίτες δεν μπορούν να συνεχίσουν να καταπιέζονται. Πρόεδρε, 5.723 ημέρες έχουν περάσει από τότε που έχει φυλακιστεί ο Νταβίτ Ιζακ. Φτάνει πια. Σας ευχαριστώ. Διαδικασία Καστιάη. Εχτώ οι ομιλητέ που είναι στο κατάλογο και θα τους δώσω σε όλους το λόγο. Ο κύριος Πόσπης, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ με το ψήφισμά μας. Και για τον Αντώνιο και για τον κύριο Ισάκ. Και πέραν αυτών θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για ένα από τα χειρότερα καθεστώτα παγκοσμίω. Πρόκειται για ένα καθεστώ που έχει καταπατήσει κάθε δικαίωμα κάθε θεμελιώδες δικαίωμα. Οι πολίτες της χώρας είναι σχεδόν σε κατάσταση δουλείας. Υποχρεωτική κατάταξη στον στρατό, δολοφονίες αντιφρονούντων και δημοσιογράφων. Νομίζω ότι σε αυτό το ψήφισμα θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να διακόψουμε την οικονομική ενίσχυση προς την χώρα θα χρησιμοποιήσουν οι κυβερνώντες τα χρήματα. Ποτέ δεν τα πάρει ο κόσμος. Επομένως δεν πρόκειται μόνο για αυτούς τους δύο κρατούμε συνείδηση, πρόκειται για ολόκληρο το λαό που υποφέρει. Η Άννα Γκόμες για ένα λεπτό είναι η επόμενη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ιζάκ είναι ένας από τους χιλιάδες Πρόκειται για τις ε, διαμαρτυρίες που έγιναν. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα αυτό, το ευρωπαϊκό ε, λαό υπόκειται σε τρομοκρατικές τέτοιες επιθέσεις και δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι λαμβάνονται τέτοια μέτρα σε ό,τι αφορά και την ε, Ερυθρέα και αυτά που συμβαίνουν εκεί χιλιάδες εκατομμύρια χωρίς ερεσιμότητα για να αντισταθούμε στην ροή τη μεταναστευτική. Αυτό δεν είναι μόνο σπατάλη των ε, πόρων. Είναι προδοσία. Προδίδουμε την εξωτερική μας πολιτική και αυτό δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα είχε στη δημοκρατική μετάβαση στην Ερυθρέα. Ευχαριστώ. Ο κ. Μότση Μαριά. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η κατάσταση στην Ερυθρέα είναι πλέον εκτό ελέγχου λόγω των πολιτικών διώξεων που κάνει το καθεστώς αλλά και λόγω της απεριόριστης αναγκαστικής στρατιωτικής θητείας. έτσι πάνω από 400.000 άτομα ή το 9% του πληθυσμού της χώρας έχει φύγει άρον άρον από την ερυθρέα αυξάνοντας τις προσφυγικές ροές προς την ευρώπη. η σεξουαλική βία είναι στην ημερήσια διάταξη όχι μόνο κατά των γυναικών αλλά και στα στρατόπεδα εκπαίδευσης ταυτόχρονα το καθεστώς ολοκληρώνει τον έλεγχό του κατά του πληθυσμού επιβάλλοντας φόρο εισοδήματος ομογενών 2%. θύματα του καθεστώτος είναι ο αμπούν αντώνιος ο πατριάρχης της ορθόδοξης εκκλησίας της ερυθρέας της μεγαλύτερης θρησκευτικής κοινότητας που έχει τεθεί υποκράτηση από το 2007 επί δέκα χρόνια αφού αρνήθηκε να αφορήσει 3.000 μέλη της ενορίας του τα οποία αντιτάχθηκαν στην κυβέρνηση επίσης και ο ακτιβιστής νταβίτ Ισάκ και αυτός υποκράτηση. άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, κύριο Σινκέλη, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είναι μία από τις χειρότερες χώρες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα η Ερυθρέα. Το ξέρουμε αυτό τα τελευταία χρόνια. Συνέχεια έχουμε καταχρήσεις. Και δεν είναι περίεργο που φεύγει ο κόσμος από αυτή τη χώρα. 400.000 έχουν φύγει από τη χώρα τους. Ακριβώς γι' αυτό. Όσον αφορά τον Ταβιτ Τισάκ, το 2009 συνελήφθη. Είναι ακόμα ζωντανός, δεν το ξέρουμε. Η κυβέρνηση όμως οφείλει να ενημερώσει τους δικούς του. Επίσης, ο Πατριάρχης, ο Αντώνιος, ο οποίος κρατείται σε άγνωστο μέρος και δεν έχει ιατρική περίθαλψη στη διάθεσή του. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να μην δίνουμε χρήματα στην Ερυθρέα. Δίνουμε 200 εκατομμύρια ευρώ και νομίζω ότι θα έπρεπε να σταματήσει αυτό μέχρι να έχουμε απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Φροντζουλίτσα, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώ, κύριε Πίτροπε, δεν βλέπουμε βελτίωση όσον αφορά τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθρέα. Ακόμα και παιδιά συλλαμβάνονται και κρατούνται εντελώς αδικαιολόγητα, κάτω από πολύ σκληρέ συνθήκε. Ο Ταβίτη Σάκα στη φυλακή αποτελεί διεθνέ σύμβολο για τον αγώνα τη ελευθερία τύπου στην Ερυθρία και θα πρέπει χωρί όρου να απελευθερωθεί με όλου του κρατούμενου συνάδεση. Επίση, η άλλη περίπτωση του Αμπού Αντώνιο και αυτό ο Πατριάρχη πρέπει να ελευθερωθεί. Παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα και γίνονται διακρίσει. Όλα αυτά πρέπει να καταδικάζονται. Και κύριε Επίτροπε, είμαι κατά, όπω γνωρίζετε, ω πρόεδρο τη ομάδα εργασία να δίνουμε χρήματα στο πρόγραμμα αυτό το εθνικό για την Ερυθρέα αν δεν λυθούν αυτά τα ζητήματα, αν δεν απελευθερωθούν οι κρατούμενοι αυτοί. Ο Πατριάρχης και ο Τάβιτ ε, επίσης Σισάκ και οι άλλοι αυτοί και οι κρατούμενοι οι άλλοι δημοσιογράφοι να απελευθερωθούν. Ευχαριστώ. Ο κ. Πόλης έχει ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ που δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με όλους τους ε, προλαλήσαντες. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω για την κατάσταση στην Ερυθρέα. Η Ερυθρέα είναι ένα από τα πιο νερά κράτη στον κόσμο και παράλληλα αντιμετωπίζει από τις πιο μαζικές παραβιάσεις ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο αυτά που προτείνουμε στο ψήφισμα για να ανασταλεί δηλαδή προσωρινά η αρρωγή προς την Ερυθρέα θεωρώ ότι αποτελεί μια πολύ καλή προσέγγιση. Θα πρέπει να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε μετρήσιμα αποτελέσματα της οικονομικής μας αρρωγής. Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε οικονομική ενέσχυση όταν κανείς δεν απαντά καν στις ερωτήσεις μας. Εδώ φυσικά σήμερα συζητάμε το θέμα ε, δύο συγκεκριμένων ατόμων, αλλά υπάρχουν αμέτρητοι άλλοι, ανώνυμοι που υποφέρουν από ένα καθεστώς που ουσιαστικά χρησιμοποιεί ένα δέκατο των πολιτών του για στρατιώτες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Κύριε Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο λαός στην Ερυθρέα περνάει έναν γουργοθά και πολύ καιρό και πρόσφατα ανεξαρτητοποιήθηκε αυτή η χώρα. Αλλά υπάρχει ένα δράμα ανθρωπιστικό και πολιτικό. Ο Ισάκ και πολλοί άλλοι και κυρίως γυναίκες υποφέρουν. Τους έχουν αποστερήσει τα θεμελιώδη δικαιώματα περνούν κατάσταση δουλείας. Μιλάμε για 400.000 ανθρώπους. Η τοπική κυβέρνηση τους έχει επιστρατεύσει και μιλούμε για 2 εκατομμύρια πληθυσμό, αλλά θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Θα πρέπει να τεθεί προϋπόθεση στην οικονομική βοήθεια ο σεβασμός των οποίων δικαιωμάτων. Οπότε θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αναδεχθούν και να υποδεχθούν τους Ερυθρέους οι οποίοι ζητούν ε, άσυλο γιατί κινδυνεύουν στη χώρα τους. Ε, ο κύριος Μπράιν Χέιζ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε μου. Δεν ευκαιρία να πούμε δύο λόγια το ψήφισμα. Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθρέα είναι πολύ σοβαρό. Αλλά τα ίδια ισχύουν και για άλλες χώρες της Αφρικής που συνεχίζουμε να ενισχύουμε. Θα πρέπει το ψήφισμα να είναι ξεκάθαρο μήνυμα. Και πιστεύω, αντίθεμα τους συνεδρούς, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις σχέσεις μας με τη χώρα που έχει μπλεχτεί σε αυτόν τον πόλεμο. Θα πρέπει όμως να κατανοηθούν οι υποχρεώσεις της χώρας. Να γίνει κατανοητό τι χρειάζονται οι πολίτες της χώρας και ίσως είμαι ο μόνος από τους αντίλους που έχει πάει τελευταίο χρόνο στην ε, χώρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να εμπλακούν περισσότερο οι συνάδελφοι για να φέρουμε την αλλαγή στην Ερυθρέα. Θα πρέπει να πλησιάσουμε αυτή τη χώρα για να αλλάξει η κατάσταση. Οι, οι δε πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάνει τη διαφορά. Βελτιώθηκε η καθημερινή ζωή. Ηλεκτρισμός, ηλιακή ενέργεια, ε, δικαιοσύνη, γενικά δυνατότητες της χώρας. Άρα είναι σημαντικό να συνεχίσουμε την χρηματοδότηση προς την Ερυθρέα, αλλά να έχουμε πιο ισορροπημένη αντιμετώπιση στην προβληματική μας. Και, τώρα... και τελευταίος ε, ο είναι ο Επιτρόπος κ. Στυλιανίδη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι συμμερίζομαι την απογοήτευσή σας για την κατάσταση στην Ερυθρέα. Και ίσως αν ήμουν ευρωβουλευτής όπως πριν, θα έλεγα φτάνει πια. Τώρα όμως, υπό τη νέα ιδιότητα, από την άλλη πλευρά, εδώ στο ημικύκλιο, Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, φυσικά και ανησυχεί για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθρέα και κυρίως για τον Πατριάρχη Αντώνιο και για τον Ταβί Τισάκ και θέλει να ισχύει και εκεί το ότι αποτελούν στοιχείο κλειδί τα ανθρώπινα και τα θεμελιώδη δικαιώματα και είναι βασικά στοιχεία της εξωτερικής μας πολιτικής. Γι' αυτό και στον πολιτικό μας διάλογο με την Ερυθρέα ξανά και ξανά το βάζουμε. Η περίπτωση του Ταβίτη Σάκ μας έχει απασχολήσει από την αρχή της αυθαίρετης σύλληψής του το Σεπτέμβριο του 2001. Συνεχίζει να κρατείται χωρίς αλλαγές χωρίς να έχει υπάρξει ε, δίκη βάση του νόμου σύμφωνα με τις ε, διεθνείς συμβάσεις που έχει συνυπογράψει η Ερυθρέα. Και αυτό συνεχίζει να μας απασχολεί όπως επίσης και η σύλληψη 10 δημοσιογράφων, κάτι στο οποίο αναφερθήκατε κι εσείς. Και επίσης και όσον αφορά τον Αμπουδε Αντώνιο, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ, τον Πατριάρχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που βρέθηκε σε κατοίκον κράτηση αλλά σε άγνωστο χώρο χωρίς να το έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία για κάποιο συγκεκριμένο παράπτωμα. Έχουμε απευθυνθεί στα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης της χώρας και στα εθνικά φόρα, ακόμα και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ήδη από το 2001. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης τακτικά κάνει δηλώσεις με τις οποίες ζητά την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατούμενων στην Ερυθρέα. Επίσης, ζητούμε τακτικά από τις αρχές της χώρας να αναλάβουν όλα τα αναγκαία βήματα προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις διεθνείς δεσμεύσεις τους, μεταξύ άλλων την ελευθερία της θρησκείας και της έκφρασης του συναρθρίζεστε κλπ. Σύμφωνα με το ψήφισμα επίσης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθρέα που εγκρίθηκε τον Ιούνιο που μας πέρασε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί με την Ερυθρέα να προσπαθεί να βελτιωθεί η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιτόπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα στηρίξει την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων που έγιναν στην Ερυθρέα βάση της έκθεσης του ΟΗΕ για την επισκόπηση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα. Συνεχίζουμε να πιέζουμε για τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθρέα και κάνουμε έκκληση στην κυβέρνηση να απελευθερώσει πολιτικούς κρατούμενους, μεταξύ άλλων βέβαια και τον Ταβίτη ΣΑΚ. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει Όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν για το πού βρίσκονται και ποια είναι η κατάσταση των ε, κρατούμενων αυτών να δημοσιοποιηθεί και να μπορούν να συναντήσουν τις οικογένειές τους και τους δικηγόρους τους, αν μη τι άλλο, για λόγους ανθρωπιστικούς. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να προάγει την ελευθερία της έκφρασης και της ε, θρησκευτική πίσης, που είναι δικαιώματα τα οποία από τα οποία πρέπει όλοι να χαίρουν, γιατί είναι οικουμενικά και έχουν να κάνουν με την ισότητα και την αρχή της μη διάκρισης. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πίτροπε και κλείνοντας την ε, συζήτηση ε, κατατεθήκαν έξι ψηφίσματα και έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση. Σήμερα το μεσημέρι θα λάβει χώρα η σχετική ψηφοφορία. Περνάμε λοιπόν στο τελευταίο σημείο της σημερινής διάταξης. Ε, έχετε διαδικαστικό να θέσετε. Κυρία Βερζία. Ναι, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να πω στον Επίτροπο ότι πολλοί εδώ τον ρωτήσαμε για τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πάνε στην Ερυθρέα. Δεν μας απάντησε όμως για τα κονδύλια αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πάνε στην Ερυθρέα. Βρίσκω ότι είναι πολύ κρίμα. Κύριε Επίτροπε, έχετε κάποια απάντηση να δώσετε για το θέμα της χρηματοδότησης. Η κυρία Βερζία το έθιξε το θέμα αυτό εκ Ευχαριστώ. Κοιτάξτε. Για, αυτή την, για αυτές τις ερωτήσεις δεν ε, μπορώ να απαντήσω τώρα. Σέβομαι το έτοιμά σας αλλά είναι πολύ δύσκολο έτσι αμέσως να απαντήσω με νούμερα. Θα προτιμούσα γραπτά να δώσω την απάντηση. Σας ευχαριστώ. Ωραία, περιμένουμε λοιπόν την απάντησή σας γραπτά.